Good morning, colleagues, Καλημέρα συνάδελφοι και σας ευχαριστώ που ήρθατε και καταφέρατε να παλέψετε με τα στοιχεία της φύσης για να φτάσετε. Έχουμε αργήσει να ξεκινήσουμε, γι' αυτό πιστεύω πως θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη ιδιαίτερα δεδομένου του περιεχομένου που έχουμε να εξετάσουμε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ανακοινώσει ε, τη Πέδου, να σα υπενθυμίσω ότι τα σημεία 6 και 7 τη ημερήσια διάταξη. Να την κοιτάξετε. Συμφωνείτε? Δεν έχει κανεί αντίρρηση. Τα σημεία 6 και 7 λοιπόν, δηλαδή για την κατάσταση ασφαλείας στη Συρία μετά την ανακοινωθή αποχώρηση των δυνάμεων των ΙΠΑ και η κατάσταση ασφάλειας στο Κωσυφοπαίδιο θα συζητηθούν μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης, η δημόσια κρόαση σχετικά με τι ε, πολιτικέ ασφάλειας θα γίνει μαζί με την Επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου δύο ε, πατώματα πάνω στην αίθουσα 3G3. Το Διευρυμένο Προεδρείο επίσης θα συνεδριάσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, την 1G3, αμέσως μετά τη δημόσια ακρόαση, περίπου στις 5.30 το απόγευμα. Σημείο 3 λοιπόν, έγκριση των πρακτικών. Έχετε κάποιο σχόλιο για τα πρακτικά της 19ης ε, και 20ης Νοεμβρίου. Όχι, υπέροχα. Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν σχόλια ή ενστάσεις, θα θεωρήσω πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Και αυτό μας περνάει στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, το ουσιαστικό δηλαδή σημείο που θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και το μέλλον της συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνικούς. Είναι πολύ επίκαιρο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ε, πρώτον, εξ ονόματος της ε, υποεπιτροπής μας, να καλωσορίσω θερμότατα τους ε, προσκεκλημένους μας, τον κύριο Γιάτσεκ Μπίλιτσα, ειδικό απασταλμένο για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση και προϊστάμενο της μονάδας ΣΕΚΠΟΛ 1, αφοπλισμός μη διάδοση και έλεγχο εξαγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Έπειτα, ο Σίκο εκ μέρου του ΝΑΤΟ και του Κέντρου Μη Διάδοση, ο κύριος Σίκο Βαντερμέρ, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Κλίνγκεντελ και ο κύριος ε, Μπρούνο Λετέ, ανώτερο επιστημονικό συνεργάτη στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των ΗΠΑ. Είναι εντυπωσιακότατο το πάνελ σήμερα και ανυπομονούμε να ακούσουμε τις ε, παρεμβάσεις σας. Επίσης, έχουμε καλέσει τον ε, επικεφαλής της ε, αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να του επιτρέψει να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί εξαιτία τη ε, γνωστή κατάσταση που επικρατεί στι ΗΠΑ, όπω γνωρίζετε. Ούτε καν ε, πληρώνεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς ένα χρόνο πριν, λοιπόν, τον Ιανουάριο του 2017, στην 30η επέτειο της υπογραφής της συνθήκης ε, αυτής, είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για ακριβώς το θέμα αυτό μετά την υπογραφή της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ανανέωσε την ε, δέσμευσή της για την τήρηση της συνθήκης και την πλήρη συμμόρφωση καθώς και έναν ανοιχτό ειλικρινή διάλογο μεταξύ της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, μπορούμε να δούμε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφόρησαν και το μέλλον της συνθήκης είναι αβέβαιο αρκετά χρόνια ε, αμοιβαίων ε, κατηγοριών πέρυσι τον, ε, κατέληξαν στον περσινό Οκτώβριο όπου ο πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε από τη συνθήκη λόγω της μη συμμόρφωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά από την ε, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ τη 4 Δεκεμβρίου, οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις τους ε, που προκύπτουν από τη συνθήκη, εκτός εάν η Ρωσία συμμορφωθεί με αυτήν μέσα σε 60 ημέρες. Το ΝΑΤΟ λοιπόν στήριξε την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και την άποψη ότι η Ρωσία παραβιάζει τη συνθήκη και έκανε έκκληση για να επιστρέψει η Ρωσική Ομοσπονδία σε κατάσταση πλήρου συμμόρφωση. Οι προσκεκλημένοι μας θα σας ενημερώσουν λεπτομερώς και γι' αυτό λοιπόν με την ιδιότητά μου Προέδρου θα σας ζητήσω να παρουσιάσετε την κατάσταση ως έχει σήμερα καθώς και τα επόμενα βήματα. Σε πρώτο στάδιο λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπελίτσα. Για να μας πείτε τις νεότερες εξελίξεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι περήφανος και πολύ ευτυχής που συμμετέχω εδώ στο πάνελ με άλλους συνομιλητές από το ΝΑΤΟ, από διεθνείς οργανώσεις εδώ στις Βρυξέλλες και όπως θα θυμάστε συζητήσαμε ακριβώ το ίδιο θέμα πριν από ένα χρόνο ακριβώς και χαίρομαι για την επιλογή των θεμάτων τη σημερινή γιατί πραγματικά είναι μια συζήτηση με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και πολύ επίκαιρη βέβαια. Σας ευχαριστώ που υπενθύμισε τα βασικά στοιχεία της συνθήκης. Τι σημαίνει συνθήκη, ποια είναι η κατάσταση σημερινή. Θα περάσω κατευθείαν στην συμπεφωνημένη ενωσιακή θέση, ευρωπαϊκή θέση, γιατί είμαστε στο εξή παράδοξο ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, συμμετέχει δεν υπογράφουν κράτος της συνθήκης, αλλά η συνθήκη αυτή ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ τα, εμάς, τα συμφέροντά μας και την ασφαλειά μας. Γι' αυτό ακριβώς συζητείται το θέμα. Ε, γίνονται δηλώσεις και διαβήματα προς τα, κράτη, τα συμβαλώμενα κράτη για την διατήρηση της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει κατά επανάληψη το λόγο για να ζητήσει από τη Ρωσία να επανέλθει στη συνθήκη, να συμμορφωθεί με τη συνθήκη και η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συνθήκη για τα πυρηνικά ενδιαμέσου ελληνικού ε, συνοψίζεται στα εξή πέντε σημεία. Πρώτον, η διατήρηση τη συνθήκη ω ε, τέτοια βιώσιμη συνθήκη είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Παρότι ούτε ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλόμενο μέρο τη συνθήκη, όλοι εποφελούνται από την προστασία και τη σταθερότητα που παρέχει. Θέλουμε επομένω να διατηρήσουμε την συνθήκη αυτή όπου ε, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφούνται. Χάρη σε αυτή τη συνθήκη, περίπου 3.000 ε, πύραυλοι με πυρηνικέ και συμβατικέ ε, πυρηνικέ κεφαλές έχουν αφαιρεθεί και καταστραφεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τη διατήρηση και τη συμμόρφωση από όλα τα μέρη της συνθήκη, με τη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δίνουν την ύψιστη σημασία στη διατήρηση μιας αποτελεσματικής συμφωνίας Διεθνού Συμφωνία για τον έλεγχο των όπλων ω βασικά στοιχεία τη ευρωπαϊκή ασφάλεια και επέκεινα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει ανησυχίε κατά επανάληψη για την ρωσική συμμόρφωση προ τη συνθήκη. Μια κατάσταση όπου ένα μέρο μόνο σέβεται τι υποχρεώσει προ τη συνθήκη δεν μπορεί να επιβιώσει. Πέρυσι, κατά την δεύτερη σύνοδο τη προπαρασκευαστική NPT τον Απρίλιο του 2018, καθώ και κατά την θεματική συζήτηση για το για τα πυρηνικά το, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2018, εμείς σε μια κοινή ε, Ευρωπαϊκή Συμφωνία είπαμε ότι ένα ε, ρωσικό πυραυλικό σύστημα δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες ό,τι αφορά ότι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα ε, δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά τη ρωσική συμμόρφωση με την συνθήκη και καλούμε τη Ρωσία να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους με ουσιαστικό και ε, διαφανή τρόπο. Η διάβρωση της συνθήκης θα έχει σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για την ασφάλεια των κρατών, των συμβαλωμένων κρατών, αλλά και της Ευρώπης, αλλά και πιθανώς και άλλων περιοχών του κόσμου. Η, τα δύο κράτη με πυρηνικά, με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, δηλαδή η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, πιστεύουν και θέλουν την διατήρηση και εμπέδωση της, του Δημερού Διαλόγου Ευρωπαϊκής ε, συγγνώμη, ε, και Ρωσίας για την ε, στρατηγική σταθερότητα. 4 Δεκεμβρίου του 2018 οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν μια αναστολή των, από τι υποχρεώσει του 60 ε, μέρε μετά τι 4 Δεκεμβρίου, εκτό και αν η Ρωσία επανέλθει σε πλήρη και μετρήσιμη συμμόρφωση ε, με βάση ε, το διεθνές ε, δίκαιο και σταματήσει παραβιάσεις. Μετά τις ανακοινώσεις αυτές, σε διμερείς συνομιλίες, ελπίζουμε οι ρωσικές αρχές να επανέλθουν σε επικοδομητικό διάλογο στην πλατφόρμα που παρέχει η συνθήκη, ούτω ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της συνθήκης καλούμε τις ρωσικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτές τις σοβαρότητες ανησυχίες με ουσιαστικό και διαφανή τρόπο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι βεβαίως θα έχουμε ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι τώρα καλύτερα είναι να συνεχίσουμε ε, με τον επόμενο μιλητή και θα πάρουμε τις ερωτήσεις μετά. Με χαρά λοιπόν δίνω το λόγο στον κύριο William Μάλβεκ ο οποίος ε, είναι ε, υπεύθυνο ε, για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των έλεγχων εξαγωγής όπλων. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. πολλές φορές μίλησα εδώ και για την συνθήκη INF και πέρσι ήμουνα εδώ. Ε, βεβαίως ε, είμαι πάντα αισιόδοξο γιατί δεν μπορεί κανείς ε, με απεσιοδοξία να αντιμετωπίσει ένα θέμα όπως είναι αυτό της, του ελέγχου των ε, όπλων κυρίω όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που δεν λειτουργεί και το σύστημα πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε γιατί είναι τόσο πολύτιμη η συνθήκη INF. Να μην λησμονούμε ότι πολλοί λησμονούν τη, την εστίαση που πρέπει να έχουμε. Η συνθήκη INF δεν ε, αποσύρει κανένα πυρηνικό όπλο, απλώς ε, αναφέρεται στους ε, πυραυλού μέσου και μικρού βεληνικούς και ελέγχει αυτήν την διαδικασία. Αυτά, αυτή η πύραυλη με τέτοιου είδους βεληνικούς πυραυλικρούς κλπ. Ε, μπορούν να φτάσουν σε γειτονικές χώρες ε, δημιουργούν ε, μεγάλη ανησυχία, προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Και γι' αυτό η σταθερότητα στο πλαίσιο αυτών των οπλικών συστημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται μία προσπάθεια ε, να βρεθούν νέα όπλα τα οποία θα είναι ε, πιο ε, σωστά και πιο ακριβή. Εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητα που έχουν οι χώρες για να δημιουργήσουν τέτοια όπλα μπορεί να έχει αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα. Στο Λονδίνο ε, ε, είχαμε ακούσει πριν από πάρα πολλά χρόνια μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, ομιλία σχετικά με τα πυρηνικά όπλα. Αυτό που, τι, προσπαθούμε να κάνουμε με τη χρήση αυτών των όπλων. Οι διαπραγματεύσεις, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πριν από πάρα πολλά χρόνια για να δούμε πώς μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση απέναντι στην Σοβιετική Ένωση και οι σύμμαχοι συμφώνησαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία και αυτή η συμφωνία προσπάθησε πρώτα να καλύψει ε, το ε, το μεγάλο βεληνικές και μετά σιγά σιγά να πάμε στο μέσο και ε, μικρό βεληνικές. Ε, και είχε, ε, η συμφωνία περιλάμβανε την ε, απόσταση πυράβλων με βελνικές από 500 μέχρι 5500 και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και δημιουργήθηκαν λοιπόν ε, οι προϋποθέσεις και συνθήκες ε, για τις ε, χώρες και οπωσδήποτε υποστηρίχθηκε η ασφάλεια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και με τον τρόπο αυτό βεβαίως μειώθηκε και η ένταση μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Το 2013 οι Ηνωμένε Πολιτείες λένε στους Ρώσους ότι έχουμε ανοιχνεύσει ότι, ε, ε ότι ε, δημιουργείται ε, πυράβλους μέσω βεληνικούς, τους τοποθετείτε σε στρατηγικά σημεία κλπ. Έγινε συζήτηση βεβαίως και στο ΝΑΤΟ και επανειλημμένα προσπάθησαν να θίξουν το θέμα απέναντι στους Ρώσους, ε, οι οποίοι και το 13 και το 15 και το 16 και το 17 απήντησαν, μα δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέτε. Καταλαβαίνετε ε, το, το Δεκέμβρη του 2017, καταλαβαίνετε το άγχος των ΗΠΑ όταν ανακαλύψαν ότι ε, κάποιοι πύραυλοι οι οποίοι υποτίθεται δεν υφίσταντο υπήρχαν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι για τέσσερα χρόνια δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι έλεγαν οι Ρώσοι και ξαφνικά με την επιφύτηση λένε «Α, ναι, τώρα ξέρουμε γιατί μιλάτε». Αυτό όμως είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Υπάρχει μια ε, ε, Special Verification Committee, αυτή η Επιτροπή λοιπόν ε, εξακρίβωσης, η οποία λειτουργεί κανονικά στα πλαίσια της συνθήκης, αλλά η οποία όμως δεν λειτουργήσε εδώ. Το Δεκέμβριο του 2017, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι Ρώσοι παραδέχτηκαν ότι έχουν τους, αυτούς τους πυράβλους, αλλά βεβαίως εντωμεταξύ είχε διαμορφωθεί στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβλήματος της μη συμμόρφωσης από πλευράς ε, της ε, Ρωσίας. Είχαμε επίσης την ίδια εποχή, δηλαδή Δεκέμβριο του 2017, μια πολύ καλή δήλωση από πλευρά ε, του ΝΑΤΟ ε, που ανεφέρεται ακριβώς ε, στην προσπάθεια των ΗΠΑ να συμμορφωθεί με την συνθήκη και την αντίθετη θέση της Ρωσίας. Και βεβαίω η Αμερικανική πλευρά εξήγησε ε, ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2014 η ρωσική πλευρά είχε προχωρήσει σε ε, σημαντικές ε, παραβιάσεις και οι σύμμαχοι τότε εξέδωσαν ένα statement, μια δήλωση ότι με λύπη διαπιστώνουμε ότι όπως διαπίστωσαν και οι Ηνωμένε Πολιτείες η Ρωσία παραβιάζει το σύστημα. Παρ' όλα αυτά όμως ε, και παρότι και οι σύμμαχοι εξέφρασαν την δυσφορία τους, ε, δεν, ε, η ρωσική πλευρά δεν άλλαξε στην ουσία στρατηγική. Μεμονωμένα και διμερώς οι σύμμαχοι μίλησαν με αξιωματούχους της Ρωσίας. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε διμερείς συζητήσεις στην Γενέβη ε, και η Ρωσία ξεκίνησε ε, με, κάποιες, ε, με κάποια αποδεκτικά για το 979 αλλά χωρίς να κάνουν κάποιο βήμα προς την συμμόρφωση είναι αγχωμένοι ακόμα οι σύμμαχοι και ασχολούνται με το θέμα γιατί πρόκειται για μια σημαντική απειλή η οποία επικρέμεται. Το ζήτημα δεν είναι εάν ε, θα γίνει πυρηνικός πόλεμος στο, όμως η δυνατότητα να χτυπηθούν ε, βασικές δομές, ε, λιμένες κλπ στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, από την άλλη πλευρά η Ευρώπη βρίσκεται κάπου ανάμεσα ε, γιατί γίνεται μια συζήτηση ότι αν χτυπήσετε εσείς από τη Ρωσία θα χτυπήσουμε στην Βόρεια Αμερική ε, και γενικώ υπάρχει μια αντιμετώπιση η οποία δεν είναι, είναι αποσταθεροποιητική οι σύμμαχοι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να κάνουν μια προσπάθεια να χτίσουν κάποιες γέφυρες και με τη Ρωσία. Μέχρι τώρα η προσπάθεια αυτή είναι ανεπιτυχής. Υπάρχει και η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την... η οποία είναι πολύ θετική και η οποία δείχνει καθαρά, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει την σταθερότητα και ότι η συνθήκη είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά πρέπει κανείς να συμμορφούνται με την συνθήκη αυτή και η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση. Εμείς λοιπόν είμαστε απολύτως ε, ε, δεσμευμένοι στην ε, δημόσια τάξη και θα θέλαμε από την πλευρά της Ρωσίας να δούμε μια καλή επικοδομητική στάση που θα βασίζεται και στις αρχές του ΑΣΑ και τις συνθήκες ειρήνης και οπωσδήποτε να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίζει την ε, ε, ευρωπαϊκή ε, ειρήνη και ασφάλεια. Θα θέλαμε ε, να δούμε προτάσεις από την ρωσική πλευρά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η στάση της Ρωσίας είναι να προσπαθεί να διαιρεί τους συμμάχους το 2007 ε, η ρωσική πλευρά είχε κάνει μια ε, πρόταση στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ε, πολλές συζητήσεις είχαν γίνει και τη δεκαετία του 90 για περιορισμούς σε οπλικά συστήματα, σε πυράβλους μέσου βεληνικούς. Ε, νομίζω ότι, ότι ε, λαμβάνοντας υπόψη πλέον ε, την γενικότερη αστάθεια σε πολλά σημεία του ε, πλανήτη ε, θα πρέπει ε, να μας οδηγήσει στο να, έχουμε, να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης το MTCR είναι πολύ σημαντικό αλλά και η συμμόρφωση με το MTCR όχι μόνο για τα πυρηνικά όπλα. και όταν μιλάμε για πυράβλους κρούς, όταν μιλάμε για βαλιστικά, όταν ε, ακόμα και ε, για χώρες οι οποίες βρίσκονται εντός ε, του βεληνικού, η συζήτηση αυτή μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον και ένα ασφαλές περιβάλλον. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι πρέπει να συνεχίσει ο διάλογος, αλλά εντωμεταξύ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Δεκέμβριο ε, είχε ανακοινωθεί μια ε, χρονική περίοδος από πλευράς των ΗΠΑ που λύγει τη Δευτέρα Φεβρουαρίου. Και έχουμε και το ρολόι των έξι μηνών που λύγει τον μήνα Αύγουστο. Ε, από το 1997 συζητάμε τα θέματα ε, και η Ρωσία έχει έξι μήνες καιρό που είναι απολύτως ικανοποιητικό διάστημα έτσι ώστε να συμμορφωθεί, έτσι ώστε ε, να, ε, να διαλύσει τα παλιά όπλα και να δεχτεί έλεγχο για τα καινούρια. Μπορεί... Πρέπει να πούμε ότι στην αρχική συνθήκη ε, ε, ε, αυτά που η καταστροφή των προβλεπωμένων όπλων έγινε μέσα σε ένα μήνα. Μπορούν να καταστρέφονται 100 πύραυλοι κρούζ κάθε μήνα και να διατηρηθούν τα, γίνουν σεβαστά τα χρονικά πλαίσια. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς με αυτήν την ελπίδα ζούμε. Ελπίζω λοιπόν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα θα δώσω με μεγάλη χαρά το λόγο στον κύριο Σίκο Βαντερμέρ, ερευνητή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Είμαι μέλος μιας ανεξάρτητης ε, Think Tank και ελπίζω λοιπόν να, μπορώ, να μπορέσω να σας δώσω μια αντικειμενική άποψη. Και νομίζω πως θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε ορισμένες μακροπρόθεσμες λύσεις που μπορεί να μην φαίνονται τόσο ρεαλιστικές τώρα, αλλά νομίζω πως είναι καλό να συζητηθούν. Ε, νομίζω πως ε, η συνθήκη δεν έχει μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης, ε, γιατί για αρκετά χρόνια τώρα και οι ΗΠΑ και η Ρωσία κατηγορούν μία την άλλη πως έχουν παραβιάσει την ε, συνθήκη. Ο πρόεδρος ε, Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου αν η Ρωσία δεν συμμορφωθεί με τη συνθήκη μέχρι τότε και την περασμένη εβδομάδα η συνάντηση που έγινε στη Γενέβη ανάμεσα στις δύο αυτές ε, χώρες ε, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Οι κατηγορίες λοιπόν και από τις δύο πλευρές ε, πρέπει να ληφθούν στα σοβαρά. Η συνθήκη θα μπορέσει να επιβιώσει μόνο αν βρεθεί μια κοινή λύση. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν αμοιβέ επιθεωρήσεις ε, για να διαπιστωθεί αν όντω υπάρχουν αυτά τα οπλικά συστήματα, γιατί μόνο με έναν τέτοιο τρόπο θα μπορούσε να ε, γίνει βιώσιμη η συνθήκη. Και για τις ε, δύο χώρες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε, να δούμε τον αυξανόμενο αριθμό των πυράβλων μέσου βελινεκούς. Η εξάπλωσή τους είναι και η αιτία για τη μειωμένη στήριξη της ε, συνθήκης. Ιδιαίτερα η Κίνα ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο για, την, ε, για τις εξελίξεις αυτές. Η πύραυλοι μέσου ε, και η κατασκευή του τόσο από τι ΗΠΑ όσο και από τη Ρωσία επιφέρουν αυξανόμενου κινδύνου αστάθειες ε, και ανασφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάρρευση της ε, συνθήκης θα έχει επιπτώσεις και σε άλλες συμφωνίες για τον έλεγχο των, ε, της διάδοσης όπλων ιδιαίτερα για τη συνθήκη μη διάδοσης τι μπορεί όμω τώρα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να καταβάλει μια τελευταία διπλωματική προσπάθεια για να διασωθεί η συνθήκη, για παράδειγμα εξετάζοντας διάφορους τρόπους ε, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση μέσω των ε, επιθεωρήσεων των οπλικών ε, συστημάτων. Ε, όμως δεδομένης τη έλλειψη πολιτική βούληση και από τι δύο πλευρέ δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου σίγουροι για τι ε, πιθανότητε επιτυχίας αυτού του σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο Β για το τι θα γίνει σε περίπτωση που μετά τι 2 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από τη συνθήκη. Ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καταρχά, οι Ευρωπαίοι ηγέτε θα ε, μπορούσαν να εκφράσουν έντονα την ε, ανησυχία τους ε, για το μέλλον της συνθήκης. Θα μπορούσαν να παροτρύνουν και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ε, δεδομένου ότι είναι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, έτσι ώστε να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις επικοδομητικές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια νέα βελτιωμένη συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών όπλων θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνδράμει ενεργά σε νέες πρωτοβουλίες για ε, ενίσχυση και αναδιοργάνωση των ε, επιθεωρήσεων αυτών. Η πρόκληση βέβαια θα είναι να πιστούν οι δύο αυτές οι ε, υπερδυνάμεις, αλλά και να μην παραγνωρίζεται ο ρόλος της ε, Κίνας. Η ασφάλεια θα μπορεί να επιτευχθεί και θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς ε, να υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης. Επίσης, Χρειάζονται ανανεωμένες προσπάθειες για να οδηγηθούμε σε μια νέα συμφωνία ελέγχου γλυκών συστημάτων. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα εύκολα, δηλαδή διάφορα μέτρα μείωσης του κινδύνου, ε, διάφορα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις ε, και κακή επικοινωνία. Επίσης, ε, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να εμπεριέχουν μια διαχείριση των ε, επιπτώσεων και επίσης ε, να εξεταστεί το ε, ενδεχόμενο της ανάπτυξης γεωγραφικών δικτύων ελέγχου. Επίσης, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε επίσης το ενδεχόμενο λεπτομερέστερων ελέγχων ε, στις ε, περιοχές όπου κατασκευάζονται και είναι σταθμευμένα πυρηνικά όπλα. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει στο ε, μελλοντικά. Τέλος, είναι αναγκαία η ύπαρξη εμπειρογνωμοσύνης οι ειδικοί εμπειρογνώμονες ε, των έλεγχο οπλικών συστημάτων ε, σπανίζουν πλέον, ιδιαίτερα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επενδύσει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης έτσι ώστε να εκπαιδευτούν νέοι ε, εμπειρογνώμονες. Επίσης, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο και να αντλήσει από τις ευέλτιστες πρακτικές όπως για παράδειγμα τον ενεργό ρόλο της στην ε, συμφωνία με το Ιράν. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσει στις ε, διπλωματικές της ε, ικανότητες. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τους συμμάχους, ιδιαίτερα με τον, με τον ΝΑΤΟ και σε γενικές γραμμές ε, θα ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μείνει ανενεργή, έτσι ώστε οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία να οδηγηθούν ε, σιγά σιγά στην αποκλιμάκωση της έντασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε την κατάσταση και ιδιαίτερα από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει. Τέλος, ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρούνο Λετέ από ε, το ερευνητή από το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που επανέρχομαι στην Επιτροπή σα ε, και που συμμετέχω σε αυτό το πρώτο πάνελ, σε αυτήν την πρώτη συζήτηση, για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα με τόσο σημαντικού συνομιλητέ θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ιστορική αναδρομή, όπως και ο Βίλιαμ. Είναι χρήσιμο να το κάνουμε αυτό για να θυμηθούμε την αξία της ε, συνθήκης ΕΝΕΦ. Η συνθήκη και η ευρωπαϊκή πυραυλική κρίση μεταξύ Μόσχας και ε, Ουάσιγκτον ε, διήρκεσε από το 1978 μέχρι το 1985. Η κρίση η πυραυλική κλίση έφτασε σε τέτοια επίπεδα, κλιμακώθηκε τόσο πολύ, που όταν υπογράφτηκε το 87 η συνθήκη INF, περίπου 3.000 ε, σοβιετικοί και αμερικανικοί ε, πύραυλοι ενδιάμεσου βελληνικούς είχαν αναπτυχθεί πάνω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ήδη. Θα ήθελα, ήθελα να ξεκινήσω μια ιστορική αναδρομή, γιατί είναι εντυπωσιακό το, να θυμηθούμε το τι παίζεται εδώ. Και ενώ ε, οι, Αμερικανοί, οι και οι Ρώσοι ε, έλεγξαν λίγο τα όπλα τους ε, και ενώ τώρα παίζουν λιγάκι με τη συνθήκη, αυτό σημαίνει, σημαίνει αυτό για τη δική μας ασφάλεια. Εάν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι αναπτύξουν εκ νέου αυτά τα όπλα και πεθάνει η Συμφωνία ΕΝΕΦ, εμείς είμαστε στο στόχαστρο. Για μας τους ε, Ευρωπαίους ε, η στρατηγική σημασία της συνθήκης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ή θα ξεφορτωθούμε τα όπλα ή θα μας έχουν στο στόχαστρο εμάς. Νομίζω ότι μόνο μία πολιτική επιλογή έχει η Ευρώπη. Είναι να πιέσει τους Αμερικανούς και τους Ρώσους να μπουν σε έλεγχο των όπλων και συνεχεία στον αφοπλισμό. Μπορεί να διασωθεί η συνθήκη. Πρέπει να συμφωνήσω με τον συνάδελφο ε, και να εκφράσω σκεπτικισμό και απεσιοδοξία. Δεν είμαι τόσο ενθουσιώδη για το αποτέλεσμα της επόμενη εβδομάδας. Παρά τις ε, ευγενεί προσπάθειες ε, του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών που πήγε στη Μόσχα και μίλησε με τον ομόλογό του, πώς θα σωθεί μια συνθήκη που κανείς δεν θέλει να διασώσει. Ας βάλουμε κάποια στοιχεία λοιπόν στο τραπέζι. α δούμε τους ρώσου καταρχάς. Καταρχά δεν υπάρχει στρατηγική αξία ε, για τα ρωσικά συμφέροντα να για να διαφυλάξουν τη συνθήκη ΑΕΝΕΦ. Οι Ρώσοι για μία δεκαετία περίπου ξοδεύουν μεγάλα ποσά για να αναπτύξουν ε, συστήματα πυραυλικά cruise και σήμερα έχουν αναπτύξει δύο SS8 μονάδες πυράβλους κοντά στο Ιουκατόνιμπεργκ και άλλη μία μονάδα στο Καπούστιντζαρ, στην, ε, στην Κασπία θάλασσα. Ε, η χρήση των πυράβλων ε, ενδιάμεσου βεληνικού τα, όπως τα είπε και ο Βίλιαμ, συμπεριλαμβάνεται στα τακτικά μέτρα των Ρώσων με ε, υβριδικές, πυραυλικές και υβριδικές, υβριδικά όπλα. Αλλά φοβούνται κυρίως την ανάπτυξη πυραυλική άμυνας των Αμερικανών εδώ στην Ευρώπη και στην Ασία ε, και μπορεί να υποσκάψει την ε, ρωσική ικανότητα για το δεύτερο χτύπημα μακροπρόθεσμα. Και επομένως η Ρωσία ε, μπορεί να είναι ανοιχτή σε εκφοβισμό. Θέλει λοιπόν η Ρωσία να εξαλείψει την θέση ε, το πλεονέκτημα πούμε, των Αμερικανών. Επομένως είναι ε, κατά των υπολογισμών. Ας δούμε τους ε, Αμερικανούς οι οποίοι συμμορφώνονταν με την INF, είναι αναμφίβολο, αλλά είναι όλο και πιο περιφερειακή ως προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Η, η σημερινή κυβέρνηση έχει αντιστρέψει την προσπάθεια του Ομπάμα. Το Φεβρουάριο του 2018 ε, έχουν ξαναβάλει, ε, έγινε η επιλογή να ξαναβάλουν ε, πυρηνικές κεφαλές σε πυρηνικά υποβρύχια. Επίσης στη Ρουμανία έχουν εκτοξευτήρες, ε, τους εκτοξευτήρες MK41, αμυντικού χαρακτήρα σίγουρα, όμως τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα ε, και εναντίον των Ρώσων. Και αυτό αναφέρεται στην ε, αναθεώρηση που έγινε για τα πυρηνικά του Φεβρουαρίου του 2018 από τους Αμερικανούς. Είναι μια νέα κούρσα ε, και αυτή ε, η κούρσα θα πλήξει την ασφάλεια των Ευρωπαίων και της Ασίας, αλλά όχι των Αμερικανών. Επομένως, το κόστος για τους Αμερικανούς είναι περιορισμένο από το θάνατο της συνθήκης. Μιλήσαμε λιγάκι για την Κίνα, αλλά θα ήθελα να σας πω δύο-τρία πράγματα ακόμα η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να απελευθερωθούν από τα δεσμά της ε, συνθήκης γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν ε, στην Νότιο-Ανατολική Ασία νέες δυνάμεις, κυρίως το πυρηνικό δυναμικό και οπλοστάσιο της Κίνας έχει ε, αναπτυχθεί και αυτό το δυναμικό μπορεί να αποτρέψει του Ρώσου και του Αμερικάνου από τη δυνατότητα παρέμβαση στην περιοχή. Βεβαίω, η Κίνα επίση είναι πρόβλημα το γεγονό ότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρο μέρος στην INF, άρα μπορεί να αναπτύξει ενδιάμεσου πυράβλου η Κίνα. Και αυτό το ξέρουν ε, και θα θεωρούν στρατηγικό μειονέκτημα οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι. Ο πρόεδρος Τραμπ κατ' επανάληψη έχει πει ότι θα αποσυρθεί από την ΕΝΕΦ και το έχει βάλει σε μια ε, γενικότερη ε, σε ένα αγώνα ας πούμε, που έχει η Αμερική απέναντι στην Κίνα και στη Ρωσία. Ε, τώρα, ε, σε μια νέα τάξη θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο η συνθήκη ΕΝΕΦ. Είμαι σκεπτικιστής. Το 2007 ε, έγινε μια κοινή προσπάθεια ε, διμερής ε, να γίνει πολυ, πολυμερής ο χαρακτήρας συνθήκης INF απέτυχε. Ε, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ε, έχει αντιδράσει πολύ έντονα εναντίον ε, κάποιων δηλώσεων πρόσφατων. Α, ε, δηλώσεων πρόσφατων. Εάν η Κίνα έμπαινε στην ΑΕΝΕΦ ως συμβαλόμενο μέρος, περίπου το 90% των 1.600 πυράβλων ε, κρούς που έχουν οι Κινέζοι θα πρέπει να καταστραφούν γιατί ακριβώς καλύπτονται από το βεληνικές προβλέψεις συνθήκη INF. Ε, με μια τριμερή ας πούμε, ε, συνθήκη INF η Κίνα θα χάνει σχεδόν όλο το πυρηνικό της δυναμικό για περιφερειακή παρέμβαση. Δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τη στρατηγική της για να ε, καλύψει την Ανατολική και Νότια θάλασσά της από οποιαδήποτε παρέμβαση ας πούμε. Και για να κλείσω σιγά σιγά, τώρα, τι θα κάνουμε μετά το θάνατο της ε, συνθήκης ΑΕΝΕΦ, ποια είναι τα σενάρια για την Ευρώπη, για το μέλλον. Υπάρχουν τρία σενάρια για την Ευρώπη. Είτε θα είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη και θα επιλέξουμε να αναπτύξουμε και εμείς τα δικά μας όπλα απέναντι στην Ρωσία. Θα επιστρέψουμε στην κατάσταση του 79. Φανταστείτε, ας πούμε, τότε τις ε, την, τις αναταραχές της, ε, διαδηλώσεις, ε, τα κοινωνικά προβλήματα κτλ. Ε, το κόστος στρατιωτικό, οικονομικό κτλ. Αν εμείς δεν θέλουμε πυράβλους στην Ήπειρο, πάλι Ενωμένη Ευρώπη, αλλά είμαστε κατά, το, και ψάξουμε άλλες λύσεις με τους διεθνείς μας εταίρους. Φυσικά, αυτό θα έχει κάποιο κόστος για τις διατλαντικές σχέσεις μας που έχουν ήδη ποστεί εντάσεις και δεν θα εμποδίσει τους Ρώσους τους ή άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν και να αναπτύξουν το πυραυλικό του σύστημα. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. Ίσως θα υπάρξει μια ε, συμμαχία ε, κρατών μελών που θα δεχτούν πυράβλους ε, κρούς ε, στο, στην Ήπειρό μα, αλλά αυτό έχει το δυναμικό να διασπάσει την ε, Ατλαντική Συμμαχία. Καμία δεν είναι λύση που, που είναι ιδανική, α πούμε, αλλά είμαστε σταυροδρόμοι και πρέπει να επιλέξουμε, γιατί ό,τι επιλέξουμε θα έχει συνέπειε τουλάχιστον για, τις επόμενες, την επόμενη γενιά. Σας ενθαρρύνω όλους, λοιπόν, να κοιτάξετε αυτό το θέμα πολύ προσεκτικά, να το συζητήσετε και ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε σε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ακούσαμε και μία αξιολόγηση και μία εκτίμηση λιγότερο αισιόδοξη. Εν πάση περιπτώσει Τώρα ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις, σίγουρα θα λάβετε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Μια, ένα πρώτο γύρο συζητήσεων. Να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσω γερμανικά. Ο κύριος Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Διότι πιστεύω πως ε, αυτή η έκθεση γεγονότων, αριθμών, είναι πραγματικά πολύ σημαντική και αδιαμφισβήτητη και πραγματικά λυπάμαι ε, για αυτά που άκουσα. Ε, με λυπεί το γεγονός ότι το μέλλον της συνθήκης είναι μάλλον ζωφερό και θεωρώ πως θα έπρεπε επιτέλους και ε, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί σαφές ότι είναι προς το συμφέρον όλων να ε, σώσουμε την ε, συνθήκη και θα πρέπει να μην αποσυνδεθούμε από τους στόχους του ΝΑΤΟ και να μην υποκύπτουμε στις πιέσεις της Ρωσίας. Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει εκ νέου μια κατηγορία απαγορευμένων μέχρι τώρα όπλων. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Και αυτό έχει ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί το 1976-1977. Αναφέρατε κι εσείς ε, τον ε, Χέλμουτ Σμιτ, ο οποίος ε, είπε ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε να απαντήσουμε κι εμείς με αντίστοιχες πράξεις, όμως αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας. Και το καλύτερο θα ήταν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και θα δούμε τι θα γίνει στην ε, συνέχεια. Οι τρεις επιλογές τις οποίες αναφέρατε είναι φυσικά επιλογές που δεν είναι ευχάριστες. Η πρώτη επιλογή τουλάχιστον όταν ε, δηλαδή αναδρομικά μπορούμε να πούμε ότι τελικά ναι, το 1976-77 καλώς πράξαμε διότι οδηγηθήκαμε ε, σε αυτήν την συνθήκη και οι ηγέτες της τότε Σοβιετικής Ένωσης είχαν ε, πράξει τελικά το σωστό όπως αποδείχθηκε. Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε όμως ε, για τον Πούτιν και δεν ξέρω εάν μπορούμε να συγκρίνουμε την τότε κατάσταση με την τώρα και ε, βάσει αυτού να πράξουμε. διότι είμαι σίγουρος πως δεν θα επαναληφθεί η ιστορία ακριβώς όπως ε, τότε. Όμως θεωρώ πως θα έπρεπε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με τον έλεγχο της ε, ε, διάδοσης οπλικών συστημάτων, να γίνουν συνομιλίες, να είμαστε μεσίτες αυτών των διαπραγματεύσεων και συνομιλιών έτσι ώστε να οδηγηθούμε προς μια λύση. Έχω μια ερώτηση. Εάν η Αμερική θεωρεί πως ε, η Ρωσία θα μπορούσε να κατευθύνει τους ε, πυράβλους μεσοφελληνικούς ε, σε διάφορες κατευθύνσεις στον κόσμο, όχι μόνο προς τα δυτικά. Θα είχε κάποιο νόημα να ξεκινήσουμε, να, να λάβουμε μάλλον την πρωτοβουλία για μια συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βελνικούς στην Ευρώπη. Διότι μην ξεχνάτε ότι όλοι στον ίδιο πλανήτη ζούμε και η ασφάλεια είναι κοινό στόχος. Ε, θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι η ισορροπία, είναι προτιμό... η στις ε, δυνάμεις είναι προτιμότερη της ανισορροπίας. Διότι καμιά φορά, ξέρετε, όταν ε, υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για όλους. Ίσως αυτό θα ήταν καλύτερο από ε, το να πούμε να πράξουμε όπως ε, είπατε. Ή θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα, αφήστε τους. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προχωρήσει πολύ δυναμικά, όμως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, μην ξεχνάτε, είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Ρωσία, από την άλλη, ε, είναι απρόβλεπτη. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει αν στριμωχτεί ίσως θα έπρεπε να κρατήσουμε μία στάση κάπου στο μέσο, όπως ακριβώς ε, είναι και η γεωγραφική μας θέση. Και να φροντίσουμε, καταρχάς, να είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι, από την άλλη όμως ε, να μην ε, ξεχνάμε ποιος έχει εδώ παραβιάσει συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα στον κύριο Πλάσκη το, τον λόγο. Ευχαριστώ. Είναι απαραίτητη η συζήτηση αυτή για το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για μια πραγματικότητα η οποία έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα μας. Και εγώ είμαι μάλλον απεσιόδοξος και επικριτικός κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήδη βρισκόμαστε ε, στην ε, λογική της άρνησης και της αποτίναξης ε, αυτής της ε, συνθήκης συμφωνίας κλπ. Και πρέπει να έχουμε λίγο ελεύθερη σκέψη. Η λογική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας που σχετίζεται με την λογική της συμφωνίας στη δεκαετία του 80. Θυμάμαι στην τηλεόραση είδα όταν ανταλλάξανε τις, ε, ε τους, ε, ε, τις πένες, τα στυλό τα οποία ε, υπέγραψαν ο Κορμπατζόφ και ο Ρίγκαν την συμφωνία. Θυμάμαι να το βλέπω ακόμα. Εν πάση περιπτώσει η λογική πλέον αυτή έχει ξεπεραστεί. Έχουμε πλέον μια νέα στρατηγική, μια νέα κατάσταση και τώρα οι Ρώσοι λένε ότι έρχεται το ΝΑΤΟ και τους περικλεί και τους πνίγει ε, και ότι εν πάση περιπτώσει ε, αυτά που θέλα, λέγανε οι άλλοι ότι κάνει η Ρωσία και δεν τα έκανε τώρα τα κάνει το ΝΑΤΟ βλέπετε ότι η λογική έχει αλλάξει και σε ένα τέτοιο περιβάλλον βεβαίως ε, η κατάσταση ε, με τη Ρωσία έχει πλέον περίπου παγιωθεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα κάνει κάποια τρομερά βήματα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, με επιρροή σε άλλες ε, περιοχές. Καταλαβαίνω τη λογική, μπορώ να δεχτώ τη λογική σε σχέση και με την Κίνα γιατί φτάνει το πλήρωμα του χρόνου που και εκείνοι θα θέλουν τέτοιου είδους ε, ε, όπλα και καταστάσεις. Ε, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να συνδυάσουμε κάποιες από τις προτάσεις σας, αλλά φοβούμαι ότι θα είναι αναποτελεσματικές. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμείς θέλουμε τη συνέχεια της συνθήκης, ότι θέλουμε να ξεκινήσουν νέες συζητήσεις και Πέρα όμως από όλα αυτά δεν νομίζω να, ότι μπορούμε πολλά να κάνουμε και θα πρέπει να προσαρμοστούμε απλά στη νέα πραγματικότητα και να κάνουμε ό,τι ε, περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι τακτικός ε, δυνατόν έτσι ώστε να κάνουμε κάποιες μικρές, ε, κάποιες μικρές βελτιώσεις από εδώ από εκεί. Είμαι απεσιόδοξο, ζητώ συγγνώμη που εκφράζομαι τόσο απεσιόδοξο, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια. <laughs> We'll work on your optimism. <laughs> Right. I now have a long list of speakers which... Έχω ένα μακρύ κατάλογο. Λόγω και του θέματος βεβαίως αυτό δεν εκπλήσει κανέναν. Θα πάρω πρώτα τους συντονιστές, θα δώσω δηλαδή πρώτα το λόγο στους συντονιστές και μετά στους υπολείπους ευχαριστώ. Ξέρουμε πού είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε. Ακούγεται ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί η κατάσταση και ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ε, όσον αφορά τις αμοιβέ επιθεωρήσεις, οι οποίες ε, είναι απαραίτητες. Κάποιος μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτή τη συνθήκη ε, και για το κατά πόσον θα μπορούσε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση αυτής της συνθήκης και ποια θα ήταν ε, η μορφή και αν θα μπορούσε να συμπεριλάβει ας πούμε και την Κίνα. Επίσης ε, έγινε λόγος για την στρατηγική του όριμου φρούτου τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσουμε να, να, να, κόψουμε αυτά τα όρημα φρούτα. Οι διπλωματικές μας ικανότητες ποιες είναι. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητές μας ή την δύναμή μας για να επηρεάσουμε. Επίσης, είπατε ότι πρέπει να πιέσουμε τον Τραμπ και τον Πούτιν. Ναι, φυσικά. Φυσικά πρέπει να το κάνουμε, αλλά πώς μπορούμε να ε, πιέσουμε τύπους σαν αυτούς τους δύο. Και οπωσδήποτε να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πιέσουμε και την Κίνα. Η κούρσα ε, των οπλισμών δεν λύνει τίποτα. Γιατί ε, όσο περισσότερα όπλα, ε, τόσο περισσότερα ακόμα θα δημιουργούνται. Να κρατήσουμε την ε, ισορροπία, αλλά με λιγότερα, όχι με περισσότερα όπλα. Να χρησιμοποιήσουμε τη διπλωματική μας δυνότητα περισσότερο, έτσι ώστε να επιτύχουμε τον αφοπλισμό. Γιατί διαφορετικά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και οπωσδήποτε είναι εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση. Thank you. Thank you very much. Now... Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια. Και εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Βαλέρο σχετικά με την επίτευξη ισορροπίας που θα τίνει όμως προς λιγότερα και όχι ε, προς περισσότερα όπλα. Και έχω μια ερώτηση σχετικά με αυτό. Πριν από λίγες μέρες διάβασα ένα άρθρο που δημοσίευσε ο καθηγητής Θεότορ Πόστελ από το MIT σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και είπε ότι ένα κομμάτι του, ε, συστήμ, του, αμυντικού, του αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει λογισμικό ε, το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα στα, στην ε, αποτροπή επιθέσεων από όπλα μέσου βεληνικούς. Σε ένα σενάριο μιας υποθετικής απειλής τι μέτρα για τον έλεγχο των όπλων θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε, έτσι ώστε ακριβώς να επιτευχθεί μια ισορροπία δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχω τέσσερις συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο με τη σειρά. Ο κύριος Φρουνζουλίκα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Για το νέο πρωτοπόρο ρωσικό σύστημα, τι έχετε να πείτε. Λένε ότι αυτό το πυραυλικό σύστημα είναι άτρωτο ε, και δεν μπορεί να το πλήξει, να το ακυρώσει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Πώ θα επηρεάσει αυτό την όποια ισορροπία υπάρχει, που δεν υπάρχει τέλος πάντων. Επίσης, τι μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται ε, ξανά μπήκαμε σε μια κούρσα όπλων, τρομερή κούρσα, και παρόλα αυτά βασιζόμαστε ε, βασίζουμε την ασφάλειά μας ε, στο λεγόμενο MAD, δηλαδή στην αμοιβαία καταστροφή. Γιατί φαίνεται να μην υπάρχει αλλιώς επίτευξη ασφάλειας. Σε τι βασίζεται τελικά η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, η βασική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο η Γαλλία, αλλά με περιορισμένο δυναμικό θα πρέπει να βασίσουμε την ασφάλειά μας στους βασικούς μας, στο βασικό μας σύμμαχο, ο οποίος είναι σε φάση απομόνωσης, απομονωτική πολιτικής απομόνωσης. Ε, έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο που φεύγει, ε, η Ρωσία που ομφαλοσκοπεί, έχει μια δική της ε, πολιτική. Υπάρχει μια πολύ ανισόρροπη κατάσταση ό,τι αφορά την παγκόσμια ασφάλεια. Μη ισορροπημένη, εν πάση περιπτώσει. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις, αλλά... Thank you. very much. I should add that there is... Ευχαριστώ. Στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο υπάρχει ένα κίνημα αντίστασης ε, στο Brexit και εγώ ανήκω σε αυτό το κίνημα, ήθελα να το πω αυτό. Τώρα, ο επόμενος ομιλητής από την Πολωνία. Να ξεκινήσω από αυτά που είπατε εσείς, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία στο, με το κίνημα αυτό αντίστασης, παρότι δεν είναι το θέμα μας. Αλλά αν είσαστε πολύ έτσι, δραστήρια σε αυτό το κίνημα αντίστασης, κάτι μπορεί να δώσει, το ευχόμαστε. Λοιπόν, Δέκα χρόνια δουλεύει αυτή η υποεπιτροπή και συμμετέχω κι εγώ. Και σπάνια ακούμε τέτοιου τύπου πληροφορίες τόσο σημαντικές, ε, ενδιαφέρουσες διανοητικά, αλλά και επί της ουσίας. Ευχαριστούμε τους ομιλητές, πραγματικά πολύ ποιοτικοί, ποιοτικές οι σημερινές παρουσιάσεις. Τώρα, συμφωνώ με τους συναδέλφους που προηγήθηκαν και που είπαν ότι Είμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή και οποιαδήποτε έλλειψη συμφωνίας θα οδηγήσει σε τρομακτικές συνέπειες ό,τι αφορά την πολιτική και σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιλογές που θα υπάρξουν. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, γι' αυτό θα εστιάσω σε δύο πράγματα. Πρώτον, θα ήταν καταστροφή αν η Ευρώπη δεν λάμβανε στήριξη από τους Αμερικανούς στις επερχόμενες συζητήσει. Το αναφέρω αυτό γιατί όλοι ξέρουμε ότι το βασικό δυναμικό του ΝΑΤΟ βασίζεται στους Αμερικανούς. Προέρχεται από τους Αμερικανούς. Ε, μια και τα ξέρετε τόσο καλά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η αντίληψή σας, πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να ε, πετύχουν συμφωνία με τους Ρώσους ή παριστάνουν κάτι τέτοιο χωρίς πραγματική πρόθεση να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε. Και δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε για την αποτυχία των ε, διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά, μια και κάθε μέρα έρχονται νέε πληροφορίε από τις ΗΠΑ που επιβεβαιώνουν ότι η χώρα ε, είναι σε μια έτσι τροχιά απομόνωση και θέλει να απομονωθεί και να αποκοπεί από την Ευρώπη. Δεν θέλει να ασχολείται με την ασφάλεια τη Ευρώπη, δεν θέλει να είναι υπεύθυνη πια για την ασφάλεια της Ευρώπης η Αμερική. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ερώτημα. Οι συνέπειε μια τέτοια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο συμφωνώ ότι έχουμε πολλά σενάρια ως προς τις πολιτικές. Τι γίνεται όμως με τις, πολιτι... με τις στρατιωτικές συνέπειες. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου από μόνοι μας, οι Ευρωπαίοι, δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό αμυντικό σύστημα απέναντι σε αυτούς τους πυράβλους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πλήρες σύστημα και ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι πρόβλημα. Μπορούμε να φανταστούμε τις πιθανές στρατιωτικές συνέπειες για την Ευρώπη εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε πούν αυτές, αυτά τα συστήματα που έχουμε στην Πολωνία και την Ρουμανία είναι σημαντικά, αλλά είναι σημαντικά για μας και για τη δική σας ασφάλεια, δικό σας θέμα, αναλάβετε τις ευθύνες σας, ε, ή πληρώστε μας αν θέλετε να είμαστε υπεύθυνοι. ποιε θα ήταν οι συνέπειε για την Ευρώπη σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ σημαντικά αυτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φρόιντ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Θα ότι παρερχόμουν στον κύριο Πάσκου. Θα έλεγα ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος και αισιόδοξο, άρα υπερέχω, όμως κοίταξα πότε γεννήθηκε και τελικά είναι μεγαλύτερος από μένα. Δυστυχώς όμως η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι αισιόδοξο αυτές τις μέρες. Ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς και ένας από τους καταλήτες αυτής της δυσκολίας στις, ε, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ονομάζεται Donald Trump. Όμως δεν ήταν ο πρώτος που έφερε αυτές τις ε, δυσκολίες, είναι η κατάσταση παλαιότερη από εκείνον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Νομίζω πως σε λίγους ε, μήνες από τώρα θα φανεί το παρασκήνιο της ε, όλης υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή όμως ε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η στάση είναι ξεκάθαρα αντιρωσική. Διότι εφόσον εξελέγει, πήρε αυτό που ήθελε στην ουσία, οπότε δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ε, ο κύριος ε, Λετέ, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι υπάρχουν ε, εκτοξευτές πυράβλων στη Ρουμανία, εκτοξευτήρες πυράβλων στη Ρουμανία, οι οποίοι αναπτύχθηκαν εκεί προσφάτως και μπορούν να χτυπήσουν εδάφη στη Ρωσία. Αν ήμουν στη Μόσχα, αυτό θα με ανησυχούσε πάρα πολύ. Αφόσον κι εσείς ε, αναφέρετε ότι η βάση αυτή μπορεί να εκτοξεύσει πυράβλου σε ρωσικό έδαφος, ε, τότε από τη ρωσική πλευρά όταν βλέπεις ότι μια χώρα μέχρι τώρα ουδέτερη στρέφει όπλα προς τα σένα, αυτό αλλάζει την αντίληψή σου. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως πρέπει και εμείς να αλλάξουμε λίγο την οπτική γωνία, να δούμε τα πράγματα με ε, τα μάτια της άλλης πλευράς, διότι πάντα υπάρχει η άλλη όψη του νομίσματος. Και αυτό μου θυμίζει έναν τσακωμό στο προάβλιο του σχολείου. Όταν τσακώνονται δύο παιδιά, κανείς δεν ξέρει ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Αλλά το σημαντικό είναι να λυθεί το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος που έχει δει στο λόγο είναι ο κύριος Μπασίρ και έχετε μέσα στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας για την εξαιρετική τους παρουσίαση. Συγγνώμη που άργησα να έρθω επίσης. Ε, να πω τώρα ότι σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση που μόλις μας παρουσιάσατε, θα πω πως θεωρώ ότι η Ρωσία είναι βαθιά αποσταθεροποιητικός ε, παράγοντας. Δείτε τι έγινε με το Αζερβαϊτζάν και με την Αρμενία με την συμπράξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στην Αμπχαζία. Υπάρχει συνεχόμενη δράση της Ρωσίας. Εξόπλησε τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ε, τι γίνεται στην Κρυμαία, στον Ντόνμπα, στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία αναμφίβολα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Και πρέπει να συνεχίσουμε να ευθυγραμμιζόμαστε με τη στάση του ΝΑΤΟ, διότι μόνο έτσι θα αποτρέψουμε την ε, Ρωσία από το να γίνει περισσότερο επιθετική. Όλα αυτά αν το καλοσκεφτούμε, έγιναν ε, από πλευρά Ρωσία διότι δεν υπήρχε μια αποτρεπτική ε, δύναμη. Δεν υπήρχε μια αντισταθμιστική δύναμη για να μετριάσει την επιθετικότητα της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μου πρέπει να συνεχίσουμε ε, τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και να φροντίσουμε το σπίτι μας. Επίσης, να αναφερθώ λίγο στην Νότια Ασία και να πω ότι η Ινδία το 1974 έφερε τα πυρηνικά όπλα στην περιοχή πρώτη από όλους τους ε, γείτονες και ανακηρύχθηκε σε πυρηνική δύναμη. Πέρυσι αγόρασε όπλα επιθετικά αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτό είναι αναμφίβολα μια πράξη που θα αποσταθεροποιήσει περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή και θα σπρώξει το Πακιστάν ε, όλο και πιο κοντά στην Κίνα. Εάν συνεχιστεί αυτός ο εξοπλισμός της Ινδίας από τις Ηνωμένε Πολιτείες, τότε θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα σχέσης με το Πακιστάν δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ινδία να συνεχίσει αυτόν τον ε, αγώνα και αυτήν την ε, καταπιεστική συμπεριφορά στην περιοχή του Κασμίρ και όχι μόνο και στις γειτονικέ ε, χώρες. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το Πακιστάν μόνο του απέναντι σε αυτήν την επιθετική στάση της Ινδίας. Και η Κίνα μην ξεχνάτε ότι μόνο για δύο αιώνες έχασε την ιδιότητα της υπερδύναμης. Όλο το, τη, όλη την υπόλοιπη ιστορία ήταν υπερδύναμη. Γι' αυτό λοιπόν Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και ας μην ε, χάψουμε αυτό που μας ταΐζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ότι η Κίνα δεν είναι ε, υπερδύναμη. Η Κίνα φυσικά και είναι υπερδύναμη και θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Εμείς οφείλουμε να συνεργαστούμε με την ε, Κίνα και να μην αρνούμαστε τα γεγονότα, αυτό που γίνεται στο στενό της Μαλάκα για παράδειγμα. Φυσικά και είναι υπερδύναμη η Κίνα. Και εμείς οφείλουμε να ενεργούμε προς το συμφέρον μας ε, μαζί πάντα με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις, το, το φάσμα τους και τώρα θα πρέπει να απαντηθούν όμως. Έχουμε 15 λεπτά για να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι τα κεντρικά στοιχεία ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η αντίδραση ε, σε αυτήν την ε, κατάσταση. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά και την τεχνογνωσία, την επένδυση σε τεχνογνωσία που μπορούμε να οικοδομήσουμε Επίσης ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία όσον αφορά την πολυμερή ε, ανταπόκριση ε, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για διμερείς σχέσεις και διμερή κατάσταση. Τώρα η πολυμέρεια χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο ε, την ε, κατάσταση αυτή. Επίσης, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ξαναβάλουμε τους δύο κεντρικούς ενδιαφερόμενους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ενδεχομένως να βάλουμε κι άλλους στο τραπέζι αυτό. Να καλωσορίσω ε, και τον κύριο Μακάλιστερ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και, και έχουμε ε, λιγότερο χρόνο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές ε, ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά το θέμα της ιστορίας ας πούμε και του παρελθόντος της συνθήκης. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ε, το, το ιστορικό αυτής της ε, συνθήκης, δηλαδή πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε, ποια ήταν η τότε κατάσταση. Έγινε η διαπραγμάτευση ε, της συνθήκης σε μια περίοδο μεγάλης αισιοδοξία, τέλη της δεκαετίας του 90, όπου είχαν γίνει τρομερές πρόοδοι στην ασφάλεια της Ευρώπης, μείωση των οπλικών συστημάτων και εκεί εντάχθηκε και αυτή η συνθήκη διότι ξέρετε ότι βάσει αυτής ε, ε, ε, αποδομήθηκαν εκατοντάδες κεφαλές. Ο πρόεδρος Πούτιν ήδη τον Ιανουάριο του 2007 είχε δηλώσει ότι η ε, συμφωνία INF δεν συμβάλλει στην ασφάλεια της ε, Ρωσίας και έγινε μια προσπάθεια πολυμέρειας του ΕΝΕΦ μετά από αυτή τη δήλωση αυτή. Δεν είναι μονάχα λοιπόν οι εμπειρογνώμονες, ε, οι Ρώσοι και μερικές φορές και οι, οι Αμερικάνοι ε, που δεν δεσμεύονται από, το, από αυτά που αναφέρονται στη συνθήκη αλλά έγινε μια προσπάθεια λέω να γίνει ε, πιο πολυμερής ας πούμε ήδη το 2008 έγινε μια πρώτη προσπάθεια ε, οι εξελίξεις αργότερα θα πρέπει να ειδωθούν υπό αυτό το πρίσμα και με αυτό το πνεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφής και επανειλημμένα ε, αναφέρθηκε στην ε, σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην συνθήκη και στα Ηνωμένα Έθνη ενώπιον όλων των χωρών το είπε αλλά και πιο διακριτικά και τον προηγούμενο μήνα σε επίπεδο ε, συμφωνημένου κειμένου και συμφωνημένης ε, θέσης ε, από τους Υπουργούς Εξωτερικών επανέλαβαν την άποψη αυτή και αναφέρθηκε νομίζω από τον Βίλιαμ ότι την προηγούμενη εβδομάδα 15 Ιανουαρίου έγινε μια διμερής συνάντηση στην Γενέβη και υποβλήθηκε ένα ε, αμερικανικό non-paper στους Ρώσους ε, για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε συμμόρφωση καταστρέφοντας ε, τα εν λόγω οπλικά ζητήματα. Νομίζω ότι μέσα σε τρεις μέρες οι Ρώσοι απέρριψαν αυτήν την πρόταση. Λυπούμε ότι, που λέω ότι και βάσει των τελευταίων εξελίξεων ε, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε απεσιόδοξοι. Επίσης, ε, πρόσφατα έγινε και χρήση ε, χημικών ε, και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε και άλλωστε και σε υψηλό επίπεδο ε, ξανάρχισε συζήτηση για την ασφάλεια της ε, χρήσης ορισμένων όπλων και εν πάση περιπτώσει γίνεται κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η Ρωσική Ομοσπονδία να συμμορφωθεί προς τις αρχές των συνθήκων. Η πραγματογνωμοσύνη αναφέρθηκε. Ναι, μία από τις ε, πρωτοβουλίες, ίσως ε, πιο μικρή, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι η διαδικασία, το πρόγραμμα εξακρίβωσης των οπλικών συστημάτων σε συνέργεια με την Euratom. Και είναι οπωσδήποτε μία κίνηση η οποία προειδεάζει ή προετοιμάζει μελλοντικέ ε, συμφωνίες ε, αφοπλισμού. Ε, η Κίνα αποσύρθηκε βέβαια από αυτή τη διαδικασία, οπότε περιορίζεται οπωσδήποτε το εύρος μιας τέτοιας συμφωνίας, ένα οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι εκεί. Άλλη ερώτηση σχετικά με τους εκτοξευτήρες. Ίσως ο Βίλιαμ θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλβεϊ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Χαίρομαι που κάνετε τόσο ωραίες παρεμβάσεις. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν θα, μπορώσω, δεν θα μπορέσω να απαντήσω μεμονωμένα στην κάθε ερώτηση. Θα απαντήσω ομαδικά σε δέσμες ερωτήσεων. Ο κ. Βαντερμίρ έκανε μια κανή πρόταση που έκανε για, λόγο για τον έλεγχο των όπλων και επενδύσεις. Η, επενδύση η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει όχι μόνο στο, στον έλεγχο των όπλων, αλλά σε, στην πολιτική α, ασφάλειας. Η, αυτό που με σοκάρει είναι ότι μειώνουν τις... Α, διώχνει προσωπικό, ας πούμε, διευθυντές ασφαλείας κτλ. Ε, και αυτό ο έλεγχος των όπλων είναι απλώς ε, ένα εργαλείο της ασφάλειας, για την ασφάλεια. Θα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική για τον έλεγχο των όπλων, όπως λεγόταν. Ε, πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξει αυτό το εργαλείο. Να επενδύσουμε και διανοητικά ε, τι σημαίνει αποτροπή, τι σημαίνει πολιτική ασφάλεια και ο έλεγχο των όπλων, πόσο κολλάει όλα αυτά. Ε, θα πρέπει να κάνουμε επένδυση σε διανοητικό δυναμικό, α πούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα εμπειρογνώμονα μόνο για τον έλεγχο των όπλων. Θα πρέπει να υπάρχει άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν την άμυνα τη ε, χώρα σα και την Ευρώπη. Να δείτε τα διάφορα εργαλεία που έχετε μπροστά σα. Και ένα από αυτά είναι ο, διατλαντικό, ο δεσμό. Ο διατλαντικό δεσμό. Πρέπει να περάσουμε πέρα από την ε, συνθήκη. Θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα ασφαλεία ποια είναι. Συμφωνώ με πολλού από εσά που είπατε ότι αυτό ο δεσμό είναι σημαντικό. Έχουμε κοινέ αξίε. Α δούμε πέρα από το σήμερα προ το αύριο. Και τέλο, για τη Ρωσία. Ε, Πώ μπορούμε να επαναφέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για τον έλεγχο των όπλων. Ε, το είπε πεντακάθαρα. Ε, το 2007, το Μάρτιο, υπόθηκε σε ομιλία ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλυθεί αυτό το σύστημα γιατί δεν, μας, δεν είναι προ τα συμφέροντά μα. Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά αυτό υπόψη. Αλλά νομίζουμε ότι και μακροπρόθεσμα η Ρωσία ε, θέλει να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό και κάποια στιγμή θα επανέλθει ε, και θα το χρησιμοποιήσει ω εργαλείο α πούμε, για να διαμορφώσει τη σχέση. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να έχουμε ε, επενδύσεις σε προσωπικό. Ε, η Δύση προσπάθησε, ε, ειδικά στη δεκαετία του 90, ε, που άλλαξε, ας πούμε, ε, το, τον τρόπο που σκεφτόταν. Η, Ρωσία όμως δεν άλλαξε ποτέ την οτροπία της. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα το πρωτοπόρο. Ε, γι' αυτό ε, έγινε η ανάπτυξη. Τι είναι αυτό. Το 9M79. Ε, θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Και τέλος, θα πρέπει να βάλω λίγη αισιοδοξία. Η Κίνα έκανε τα δικά της μέχρι στιγμή στο διεθνές στερέωμα. Ε, πρέπει να σκεφτούν και αυτοί πώς μπορούν να συνεισφέρουν στον έλεγχο των όπλων. Ε, είναι σημαντική η δύναμη, είναι υπερδύναμη. Πρέπει να αναγνωρίσει τις ε, ευθύνες της υπερδύναμης, που δεν σημαίνει απλώς να επενδύνει σε συστήματα που αποσταθροποιούν, αλλά επενδύει και σε, στη συνεργασία για την ασφάλεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί η συνθήκη INF, να γίνει πολυμερής. Αλλά αν δείτε ε, τα όρια, ας πούμε, νομίζω ε, ότι πρέπει να βάλουμε κάποια όρια για τους ε, πυράβλους ενδιάμεσου και μεγάλου βεληνικούς. Ας δούμε ξανά την, τι είπε η Ρωσία το 2007, ας πούμε, που είπε ότι δεν θέλει να γίνει πολυμερή συνθήκη. Ας δούμε το MTCR και ας δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται όμως ε, για τη συνθήκη. Ε, και υπάρχει ένα αστείο, ε, μόνο μη, δια, μην διαταράσεις την προσπάθεια ενός ε, εχθρού σου ε, όταν κάνει λάθος. Ε, αλλά και όταν βλέπει ότι εμεί συνεχίζουμε έτσι, η Ρωσία δεν θα κάνει τίποτα. Όταν βλέπει ότι αλλάζουμε όμω, ότι επενδύουμε στην κοινή μα άμυνα και στου δεσμού μα, τότε μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι. Αλλά μέχρι να καταλάβει ότι είμαστε σοβαροί, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Επομένω, θα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά την υπόψη την άμυνά μα, να συνεργαστούμε με του διεθνεί εταίρου μα, να δούμε παντού στον κόσμο. Δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, είναι παγκόσμιο θέμα αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι εταίρου έχουμε σε όλο το πλανήτη και να ε, είμαστε πολύ πιο σοβαροί για το θέμα τη άμυνά μα. Ε, ευχαριστούμε για αυτή την πολύ δυναμική απάντηση σε αυτή την πληθώρα ερωτήσεων. Ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω πως ε, ακούστηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Στο παρελθόν δεν είχε εκδηλωθεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ε, για αυτό το θέμα, όμως βλέπω σήμερα πως ε, και η προσέλευση και οι ερωτήσεις ε, δείχνουν το αντίθετο. Θα ήθελα να εστιάσω σε κάποιες από αυτές. Να πω καταρχάς ότι ο διάλογος παραμένει ουσιώδης και πολύ σημαντικός. Χρειάζεται να βρούμε ένα κοινό τόπο, κοινό συμφέρον έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση υποφελή για όλους και η ασφάλεια είναι ένας από αυτούς τους ε, κοινούς τόπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία ε, δεν αποτελεί κίνδυνο και να δούμε επίσης ε, ότι, η, ότι τα βαλιστικά συστήματα άμυνας ίσως χρειάζονται. Πολλοί θεωρούν ότι Ακόμα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θεωρούν ότι ε, είναι σχεδόν γελίο να ανησυχούμε τόσο πολύ. Όμως ε, νομίζω πως αυτή η αντιμετώπιση είναι λανθασμένη. Το ΝΑΤΟ δέχτηκε πολλούς νέους ε, συμμάχους τα τελευταία χρόνια, αλλά θεωρώ πως μόνο όταν πάρουμε στα σοβαρά τα γεγονότα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κλιμάκωσης Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κίνα, φυσικά και η Κίνα είναι πολύ σημαντικό εταίρο στι ε, διαπραγματεύσει και στι ε, συζητήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπα ότι πρέπει να αρχίσουμε πρώτα από, το, από τα εφικτά, τα εύκολα, να πω ότι ναι, οι διαπραγματεύσει είναι κάτι τέτοιο. Αλλά τι πρέπει να κοιτάξουμε, ε, τι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στι διαπραγματεύσει. Καταρχά, μείωση του κινδύνου και μέτρα αντιμετώπιση αυτού. να θεωρήσουμε ότι είτε εκούσια είτε ακούσια ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα μέσω φελληνικού. Επίσης αναφέρθηκε και η κυβερνασφάλεια των ε, οπλικών συστημάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να βελτιώσουμε. Τώρα θα μια συνθήκη λίγο τροποποιημένη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνικού είναι μία λύση. Η Ρωσία, α πούμε, θα μπορούσε να μην έχει ε, τέτοια πυρηνικά όπλα κοντά στα σύνορα τη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό που θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι επικοδομητικές ουσιαστικές συζητήσεις. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζονται εμπειρογνώμονες, χρειάζονται, ε, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ε, να ξέρει γιατί μιλάει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα μπορούσε να επενδύσει στην ανάπτυξη τέτοιων ε, δυνατοτήτων, στην κατάρτιση εμπειρογνωμόνων μέσω, για παράδειγμα, της δημιουργίας ε, μιας ανεξάρτητης ε, ομάδας ειδικών οι οποίοι θα ελέγχουν όλες τις ε, λεπτομέρειες μιας τέτοιας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μέσου Βελληνικούς. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και καλά καταρτισμένοι για τον ενδεχόμενο διάλογο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα κάπως άτυπο φόρουμ όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Τέλος. Να πω πως ε, μπορεί να είμαι νεότερος από εσά, αλλά είμαι αισιόδοξο, ε, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε απεσιόδοξοι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και σίγουρα Κάθε άλλο παρά ιδανική είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όμως οφείλουμε να παραμείνουμε αισιόδοξοι έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να την βελτιώσουμε. Ελπίζω λοιπόν να κατάφερα να σας ε, δώσω έμπνευση για να συνεχίσουμε ε, τις προσπάθειες προς μια κατάσταση αμοιβέ αποφελή για όλους. Σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, ίσως τώρα είναι λίγο πιο αισιόδοξο ο κ. Ναι, νομίζω ότι άλλωστε ε, το πνεύμα κάνει τη νεότητα, όχι η ηλικία. Thank you, Madam Chair, and Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις ε, τις οποίες θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ε, θα εστιάσω λοιπόν την προσοχή μου στις ερωτήσεις που είχατε. Κύριε Φραντζούλη, κάνατε μια ερώτηση, θα σας απαντήσω. Οι εκτοξευτήρες οπωσδήποτε βρίσκονται στην καρδιά της διαφωνίας ε, των, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί οι εκτοξευτήρες ε, ε, αφορά τους ground launchers και αφορά την Αμερικανική ασπίδα προστασίας, θα μπορούσα μάλιστα να πω την Ατοική ασπίδα προστασίας και αυτή η εκτοξευτήρες ε, ε, ε, είναι καθαρά αμυντικού χαρακτήρα. Δεν έχουν να κάνουν με επιθετικούς πυρήνε, με τεχνικούς πυράβλους αλλά βεβαίως με κάποιες τεχνικές προσαρμογές είναι γεγονός ότι θα μπορούσαν να γίνουν και επιθετικοί πυράβλοι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει τώρα. Οι εκτοξευτήρες αυτοί επίσης συμμορφούνται προς τους κανονισμούς της συμφωνίας ε, της συνθήκης INF. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Ε, σχετικά με αυτό που λέτε ότι αν είχα απέναντί μου τέτοιους εκτοξευτήρες ε, θα προβληματιζόμουν, το κατανοώ. Αλλά ε, η ε, Ρωσία χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα αυτούς τους εκτοξευτήρες έτσι ώστε ε, να προχωρήσει σε παραβιάσεις και αυτό δεν είναι καθόλου επικοδομητικό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια στοιχεία διαφάνειας, έναν μηχανισμό ελέγχου και έγινε κάποια, ε, ε, κάποια ε, πρόταση από πλευρά των ΗΠΑ σχετικά, η οποία επιβεβαιώνεται και από τον Αμερικανό εκπρόσωπο, αλλά δυστυχώς δεν την δέχτηκε η Ρωσία. Επαναλαμβάνω, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι καθαρά αμυντικού χαρακτήρα και με κανένα τρόπο δεν αποτελούν παραβίαση της συνθήκης. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά την ισορροπία που αναφέρθηκε προηγουμένως. Κοιτάξτε, μόνο μέσω της ενότητας πώς επιτυγχάνεται ε, η ισορροπία. Ε, η ισορροπία ε, στην Ευρώπη αλλά και διατλαντικά μέσω του ΝΑΤΟ. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ωστόσο είναι γεγονός ότι αυτή η συνθήκη δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των υπολογισμών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, προς τα τέλη ε, ε, της, θητείας Μπούς και στη διάρκεια της θητείας Ομπάμα άλλαξαν κάπως οι ισορροπίες αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί για την Ευρώπη, καθόλου μάλιστα δεν εννοώ αυτό. Ωστόσο, ο, ο κύριος Πάσκου είπε προηγουμένως ότι ε, έχουμε την αίσθηση ότι ε, μεγάλες χώρες χρησιμοποιούν την Ευρώπη ε, σαν διαπραγματευτικό εργαλείο ή ότι χρησιμοποιούν την Ευρώπη σαν πεδίο μάχης. Δεν έχω τη δική σας εμπειρία κύριε Πάσκου αλλά ε, ε, πραγματικά ε, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να συζητήσουμε. Ναι, αλλά όχι να συζητήσουμε με τον τρόπο με τον οποίο συζητούμε τώρα, με διαφορετικό τρόπο πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις. Η Ευρώπη μιλάει με την Ευρώπη με το σκεπτικό ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει κάπως να σταματήσει. Όχι να σταματήσουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά το διαπραγματευτικό μας στυλ λίγο να αλλάξει. Θα πρέπει να ξανα ε, να σκεφτούμε ότι το INF ξεκίνησε μέσα από κλιμάκωση ε, των οπλισμών, μέσα από δύσκολες πολιτικές συνθήκες, μέσα από ε, προσπάθεια δύσκολης διαπραγμάτευσης ε, ίσως όμως το πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν έχουμε μία στρατηγική απέναντι στη Ρωσία, αλλά 28 στρατηγικές απέναντι στη Ρωσία. Θα επανέλθω στην ενότητα και την ισορροπία. Δεν πρόκειται να επιτύχουμε ε, ισχυρή θέση ή δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις από θέση ισχύω εάν δεν καταφέρουμε να ε, έχουμε ενωτική ε, θέση. Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο όμως με τον οποίο ε, συζητούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις ε, στις οποίες είχα την τιμή να ε, προεδρεύσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και εσάς και όλους τους ε, συναδέλφους που μας δώσατε λίγα από τον πολύτιμο χρόνο σας σήμερα το πρωί. Φυσικά και θα συνεχίσουμε όλοι να χτίζουμε το μέλλον, το αισιόδοξο μέλλον που όλοι επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ.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 Ε, συνάδελφοι, να ξέρετε πως ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας και δεδομένων των ε, πολύ σημαντικών ε, θεμάτων που έχουμε να συζητήσουμε πριν περάσουμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συνεχίσουμε και να δώσω το λόγο στον κύριο Πικούλα για να μας ενημερώσει σχετικά με την ε, αποστολή στην ε, Τουρκία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Να σας ενημερώσω εν για το τι συνέβη στην αποστολή. Καταρχάς είχαμε πάρα πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη. Η αποστολή έγινε από τις 17 19 Δεκεμβρίου στη Γαζιαντέπ και στην Άγκυρα και επίσης η αποστολή συνέπεσε με την συνάντηση JPC στην Άγκυρα. Ο στόχος ήταν να συζητήσουμε τις ε, ένοπλες σειράξεις στην περιοχή γειτονικά της Τουρκίας αλλά και τις σχέσεις Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε λίγες μέρες πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει την αποχώρηση των ε, στρατευμάτων των ΗΠΑ από την ε, Συρία και λίγο πριν την, άμε, την επίθεση της ε, Τουρκίας ε, σε Συριακό έδαφος. Η Τουρκία έχει πάνω από, υποδεχτεί πάνω από 2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες ε, κοντά στα σύνορα με την Συρία. Ιδιαίτερα στην περιοχή Κιλής υπάρχουν περισσότεροι Σύριοι πρόσφυγες από ότι Τούρκοι πίκοοι. Η Γαζιαντέπ επίσης βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες, όμως στην ε, πόλη αυτή βρίσκεται η πλειοψηφία των προσφύγων. Μετά, Κωνσταντινούπολη, η κατάσταση επιδεινώνεται ε, και οι εντάσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους ε, κατοίκους αυξάνονται. Επίσης υπάρχουν εντάσεις και μέσα στην σιακή κοινότητα. Είχαμε συναντηθεί στην αποστολή μας με εκπροσώπους της αντίστασης στην Συρία αλλά και ε, διάφορους ε, φορείς επιτόπου. Τα θέματα που συζητήθηκαν φυσικά ήταν ο πόλεμος στη Συρία, ε, πόλεμος τον οποίο περιέγραψαν ως πολύ ως έναν πόλεμο με πολλά πρόσωπα, κανένα όμως από αυτά δεν είναι καλό. Το Ιράν επίσης ανέπτυξε διάφορες δυνάμεις στην περιοχή, θεωρείται αντίπαλος της ε, Ρωσίας ε, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία της Αστάνα. Ο πόλεμος κατά του Άισις ε, μένεται ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαχητές οι οποίοι ενδέχεται να επανανεργοποιηθούν ανα πάσα στιγμή. Υπάρχουν επίσης αδιέξοδα μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Εθνών. Η αντιπροσωπεία μας λοιπόν εξέφρασε την ανησυχία της ε, σε ό,τι αφορά την ε, επιθετική ε, αποστολή ανατολικά του Εφράτη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους σύρους πολίτες και να διευκολύνουν τη μετακίνηση πληθυσμού προς τις περιοχές όπου παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, δεν είναι όμως αρκετή. Και σε ό,τι αφορά τους δωρητές υπάρχουν μεγάλοι δισταγμοί για κάποιους ε, συνομιλητές φαίνεται πως ε, οι, καθεστοτικέ εξελίξει καθεστοτικές εξελίξεις στη Συρία είναι αποτρεπτικές για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάποιοι άλλοι περιμένουν τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν δράση. Κάποιοι άλλοι επίσης περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια στρατηγική για την περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών συναντήθηκαν με μέλη ε, της Επιτροπής Άμυνας του Τουρκικού Κοινοβουλίου. Συζητήθηκαν οι διάφορες ε, βελτιώσεις, ε, βελτιώσεις εντός εισαγωγικών, διότι στην ουσία αυτό που σήμαινε είναι ότι πλέον ας πούμε, έχουν ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα χωρίς όμως να λείπουν οι διαφωνίες. Οι, σχέσεις, οι θέσεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης απέναντι στις, ε, στην ανάπτυξη της Τουρκίας ήταν επίσης ένα θέμα που συζητήθηκε. Συζητήθηκε και η απόπειρα πραξικοπήματος πριν από μερικά χρόνια στην ε, Τουρκία καθώς και η ασύμετρη στάση, αντίδραση της Τουρκίας ε, στην, ε, στην απόπειρα πραξικοπήματος. Η, συζητήθηκε επίσης η καταστολή της ελευθερίας ε, του λόγου, οι διώξεις και φυλακίσεις δημοσιογράφων και διανοούμενων και επίσης να κλείσω λέγοντας ότι η συνάδελφος Μποντήλ Βαλέρο από τους Πρασίνους συμμετείχε στην αντιπροσωπεία και η αντιπροσωπεία έλαβε πληροφορίες ε, για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και στα σύνορά με τη Συρία από πρώτο χέρι. Η σχέση μας με την Τουρκία παραμένει επιβαρημένη, μας χωρίζουν πολλά, όμως χρειάζεται να επενδύσουμε σε στρατηγικές ε, εταιρικέ σχέσεις στην ε, περιοχή αυτή, έτσι ώστε να δοθεί μία λύση στο προσφυγικό θέμα και το θέμα της ασφάλειας στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνατε μια λεπτομερή ε, ανάλυση της ε, κατάστασης και του τι έκανε η Επιτροπή Επιτόπου. Κυρία Βαλέρα, ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος ε, τα εξήγησε όλα εν λεπτομερία. Λίγα έχω να προσθέσω λοιπόν. Αλλά να πω δύο λόγια παραπάνω σχετικά με το τι έγινε στη συνάντηση με την Συριακή Αντιπολίτευση Είχαμε, είναι τρεις ε, διαφορετικές ομάδες ε, που δουλεύουν, που δρούν στην ε, Συρία και στην ουσία στην περιοχή του Αφρίν εκείνη την εποχή επιχειρούσαν βόρειο ανατολικά λοιπόν της Συρίας όπου γίνεται γίνεται προσπάθεια εκρίζωσης ε, της ε, τρομοκρατίας ε, και όχι μόνο με το ΠΚΚ αλλά και το PID και το IPG. Εντάξει, στην αρχή λέμε Βόρεια Συρία, Βορειοανατολική Συρία, μιλάμε περίπου για την περιοχή Αφρίν. Όταν μας, τους ρωτήσαμε όμως τι θέλουν να κάνουν, αναφέρθηκαν στο σύνολο του Βορρά. Όπως είπε ο συνάδελφος ήδη, εμείς είχαμε την αίσθηση ότι θα γινόταν εισβολή σε ορισμένες ε, ώρες. Τελικά δεν έγινε και χαίρομαι γιατί ούτε τότε έγινε ούτε τώρα ακόμη έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ε, να δουλέψουμε έτσι ώστε να μην αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί και εάν αποσυρθεί η το, οι Ηνωμένες Πολιτείες αν αποσυρθούν από την Συρία θα είναι πολύ πιο εύκολο να, κάνει εισβολή η Τουρκία. Και βεβαίως γνωρίζουμε και κάποιοι από την ΝΤΑΕΣ έχουν πάει στις ομάδες των, And, uh, there, all... των ανταρτών. Γιατί αν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση θα είναι πραγματικά καταστροφικό σενάριο. Κάτι άλλο. Θέλω να πω, ναι, ε, ε, μας υποδέχθηκαν με μεγάλη αγένεια, πρέπει να πω. Και αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Όταν πηγαίνει σε μια χώρα προσπαθούν να συμπεριφερθούν σωστά και να έχουν διπλωματική στάση. Αυτό όμως δεν συνέβη ούτε στην Επιτροπή Άμυνας, ούτε στο ε, Υπουργείο με τον Υπουργό ε, Άμυνας στο ΖΕΠΙΣ ήταν λίγο πιο ε, ευγενείς, αλλά παρόλα αυτά συνέχεια μας έλεγαν ότι θέλουν την υποστήριξή μας ε, στην εισβολή στη Βόρεια Συρία, γιατί είμαστε από την ίδια πλευρά, πολεμώντας την τρομοκρατία. Είναι κάτι που έχουμε από κοινού. Ναι, βαχόμαστε ε, κατά της τρομοκρατίας μαζί. Άρα μας έλεγαν ότι θα πρέπει να είμαστε μαζί τους σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι το μήνυμα που πήραμε από την Τουρκία. Παντού, όπου και αν πήγαμε. Ευχαριστώ. Thank Πρόεδρος, ναι, ναι, πραγματικά ήταν σημαντική αυτή η επίσκεψη. Ζητώ συγγνώμη τον κύριο Μακάλιστερ γιατί ε, καθυστερούμε το επόμενο σημείο στην αποκοινού, την αποκοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δηλαδή, ναι, ήταν πολύ σημαντική η αναφορά που μας κάνατε. Γι' αυτό θα θέλαμε ε, να μας τη δώσετε για γραπτά και για να μπορέσουμε να την στείλουμε και σε όλους τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, με μεγάλη ταπεινότητα αλλά και κάποια μηχανία, στρέφομαι προς τον Πρόεδρο ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε και θα του παραχωρήσω τη θέση μου στην Προεδρία ε, και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πίκουλα και κυρία ε, Βαλέρα για την ε, αναφορά που κάνατε σχετικά με την επίσκεψή σας.